Ε, αποστέλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό στην Επιτροπή Νομική. Ε, τρεις γραπτές ε, δηλώσεις, καταρχήν η 15-2015, σχετικά με την πρόσβαση στον τουρισμό από τον κύριο Γκάσπαρα και, και άλλα 10 μέλη συγκεντρώσε 387 υπογραφές. Υπάρχει και η δήλωση 17-2015 για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού από την κυρία Childers και 9 ακόμη μέλη. Συγκεντρώθηκαν 394 υπογραφές. Και η δήλωση 18 του 2015 για τον αυτισμό υποβληθής από τον κύριο Καπούτο και, Καπούτο και 30 ακόμα μέλη συγκέντρωσε 418 υπογραφές. Αυτές με τα ονόματα των ε, υπογραφώντων ε, θα σταλούν ε, στους παραλήπτες και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά σήμερα με βάση το άρθρο 231.4 ε, των διορθωτικών ε, εγκρίνονται τα, πρακτικά, τα διορθωτικά πρακτικά των αρμοδίων επιτροπών. υπάρχουν στην δικτυακή